Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σα παρακαλώ να καθίσετε για να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Η πρώτη έκθεση είναι έκθεση κυρία Μετσόλα, ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μία ψηφοφορία ονομαστική και ενιαία αρχίζει τώρα.